και τη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο τίτλος θα ανακοινωθεί στα πρακτικά της συνεδρίασης. Η τρίμηνη διορία που διαθέτει το Κοινοβούλιο για να ε, γνωμοδοτήσει αρχίζει αύριο 19 Σεπτεμβρίου 2014. Τα πρακτικά της συνεδρίασής μας θα υποβληθούν προς έγκριση στην αρχή της επόμενης συνόδου και αν δεν έχετε αντιρρήσεις ε, θα διαβιβάσω τα ψηφίσματα που εγκρίναμε στους αρμοδίους φορείς και στα πρόσωπα που αναφέρονται. Διακοπή της ε, Συνόδου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και λήξη συνεδρίας. Ευχαριστώ.